Στην ημερήσια διάταξη έχουμε τώρα τη συζήτηση, την κοινή συζήτηση όσον αφορά την Ινδονησία. Σύσταση Ζαντόρ για την εθελοντική συμφωνία εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Ινδονησία σχετικά με την επιβολή δασική νομοθεσία, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλία και των διαφόρων προϊόντων που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε και τη δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Θεωρητική Συμφωνία Εταιρική Σχέση Ευρωπαϊκή Ενώση Ενδουσία σχετικά με την υποβολή τη δασική νομοθεσία, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλία και των προϊόντων αυτή που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνω το λόγο για τέσσερα λεπτά στον εισηγητή, τον κύριο Ζαντό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, καλησπέρα κύριε Επίτροπε, καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι και ευχαριστώ που είστε εδώ αργά σήμερα το βράδυ για να συζητήσουμε σημαντικό θέμα. Ήδη εξέφρασα την ικανοποίησή μου για την όλη διαδικασία επεξεργασία που οδήγησε σε ομόφωνη ψηφοφορία στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω προφανώς τους κοιόδη συγητές, κυρίες Κόστιγκερ και Μπέρντερ, τον κύριο Μάρτιν, Ζαραντίν και Μέρφυ για τη συνεργασία τους και να επενθυμίσω ότι ήταν ομόφωνη η ψηφοφορία όσον αφορά το ψήφισμα διότι θεωρούμε στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ότι αυτό είναι σημαντικότατο ζήτημα. Υπήρχε βούληση να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο όσον αφορά τη σοβαρότητα του έργου μας και τις φιλοδοξίες που έχουμε όσον αφορά την εξακρίβωση και την πλαισίωση του εμπορίου ξυλίας και προϊόντων ξυλίας και πόσο σοβαρά βλέπαμε αυτού του είδους τη συμφωνία με την Ινδονησία και προηγουμένως με κάποιες αφρικανικές χώρες. Ήταν η ευκαιρία για μένα λοιπόν να ευχαριστήσω και τις αρχές της Ινδονησίας, την πρεσβεία, όλους τους φορείς που μας επέτρεψαν να εργαστούμε. Όπως ε, είπα, θεωρήσαμε ότι το θέμα αυτό ήταν σοβαρό, συνεπώς θελήσαμε να, καλύψουμε τους περισσότερους φορείς Ινδονήσιους και Ευρωπαίους να έρθουμε σε επαφή με τους εμπλεκόμενους φορείς για να κάνουμε τις καλύτερες συστάσεις ούτως ώστε η συμφωνία που θέλουμε να είναι η καλύτερη δυνατή και πάνω απ' όλα να εγγυάται ότι η ξυλία και τα προϊόντα ξυλίας που θα εισάγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανταποκρίνονται σε κριτήρια βιωσιμότητας προφανώς. Αυτή η συμφωνία εθελοντική εταιρικής συνεργασίας με την Ινδονησία είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι τα δάση τη Ινδονησίας είναι τεράστια, είναι δάση, τα τρία μεγάλα δάση, του, μέσα στα τρία μεγάλα δάση του κόσμου και είναι μεγάλο διακύβευμα και για το κλίμα, το ξέρουμε αυτό, διακύβευμα βασικό για τη βιοπικιλότητα και προφανώς είναι βασικό διακύβευμα από την έποψη των πληθυσμών που θέλουν να ζουν στο δάσος ή ζουν από τα δάση. Είναι μια συμφωνία σημαντική διότι γνωρίζουμε τη σημασία που έχει το εμπόριο ξυλία στην Ινδονησία και με προορισμό την Ασία. Είναι σημαντικό λοιπόν οι διάφορες άδειες που θα χορηγούνται να μπορούν με κάποιο τρόπο να επιβάλλουν σωστά κριτήρια όσον αφορά τις εξαγωγές της Ινδονησίας. Κυρίως όσον αφορά το εμπόριο ξυλίας. Προφανώς, από τη στιγμή που το Κοινοβούλιο, αν έτσι πάει η ψηφοφορία αύριο, συμφωνήσει, αν συμφωνήσει το Κοινοβούλιο, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει βάσει της αξιολογήσεώς της αν το σύστημα επαλήθευσης της νομιμότητας της ξυλίας είναι σωστό και ανταποκρίνεται στα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και παρά τις προσπάθειες που έκανε η Ινδονησιακή κυβέρνηση, ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμα ανεπάρκειες. Υπάρχουν ανεπάρκειες που θέλαμε να αποδείξουμε όσον αφορά την νομοθεσία. Ανεπάρκεια όσον αφορά το επίπεδο επαλήθευσης όσον αφορά ξυλία και προϊόντα ξυλίας που προέρχονται από τη μετατροπή των δασών ε, που αλλάζει η καλλιέργεια για λόγους γεωργίας ή παραγωγή ε, φινικέλεου. Και δεν υπάρχουν σωστοί έλεγχοι όσον αφορά τη διαδικασία διοδότησης. Και ξέρουμε ότι η διαδικασία επαλήθευσης νομιμότητας δεν κάνει διάκριση μεταξύ προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί και εκείνων που δεν έχουν πιστοποιηθεί στον όλο κλάδο. Ε, γίνονται προσπάθειες, βλέπουμε χες Ινδονησίας και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του τομέα στην Ινδονησία, κοινωνία των πολιτών, ότι καταβάλουν προσπάθειες, αλλά εφόσον θα είναι η μοναδική φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εκφράσει ε, με μεγάλη ισχύ τι περιμένει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γι' αυτό θελήσαμε να κινηθούμε και το τρόπο εδώ. Και ο στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ο εξή. Η συμφωνία θελοντική εταιρική συμφωνία και οι άδειε που θα δοθούν να ανταποκρίνονται στου στόχου τη προστασία του κλίματο, προστασία τη βιοπικιλότητα, εξασφαλίζοντα προφανώ και τη βιώσιμη ανάπτυξη τη Ινδονησία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Επίτροπος ο κ. Ποτότσνικ έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, Καλό βράδυ σε όλους. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σε σημαντικό σταθμό του ταξιδιού που έχουμε ξεκινήσει με την Ινδονησία. Το ταξίδι αυτό ξεκίνησε το 2006 με το ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων ε, πάνω στην ε, εθελοντική συμφωνία συνεργασίας FLECT. Ε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή Γιάννικ Ζαντό καθώς και τους σκιώδεις οι για τη δουλειά που έχει γίνει. Την εκτιμώ ιδιαίτερα. Όπως και με όλες τις διαπραγματεύσεις, το τελικό αποτέλεσμα είναι συμβιβασμός ανάμεσα στα διάφορα συμβέροντα και ε, αποτελεί και συμβιβασμό ανάμεσα στις ελπίδες και, τον, και την πραγματικότητα. Πιστεύουμε ότι είναι καλό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό ήταν χαρά και τιμή μου να εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την υπογραφή της ε, Εθελοντικής Συμφωνίας Εταιρικής ε, Σχέσης με την Ινδονησία τον Σεπτέμβριο πέρσι. Χαίρομαι που η Επιτροπή ψήφισε ομόφωνα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος ώστε ε, να έχουμε την συγκατάθεση του Κοινοβουλίου ε, για τη σύναψη της συμφωνίας αυτής ε, και προσλέπω στην αυριανή ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Όσον αφορά τώρα το ψήφισμα και την όλη συζήτηση, θα ήθελα να τονίσω το θέμα της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην παρακολούθηση της εφαρμογής του ε, Συστήματος Διασφάλισης Νομιμότητας της Ξυλίας, ε, ε, το οποίο αναφέρεται σε διάφορες παραγράφους του ψηφίσματος. Η αναγνώριση της κοινωνίας των πολιτών είναι σημαντική για να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία του συστήματος. Για να είναι αποτελεσματικό όμως χρειάζεται να γίνει οικοδόμηση δυναμικού, να υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες καθώς και πρόσβαση στις δασικές περιοχές, καθώς και και σε παρατηρητές. Σημειώνουμε τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο αυτό. Κάποιες ε, ανησυχίες ε, που αναφέρθηκαν όπως είναι τα δικαιώματα έγκυας ιδιοκτησίας ξεπερνούν τα όρια των όσων μπορεί να κάνει η Κομισιόν ε, στο πλαίσιο της θελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης και θα απαιτήσουν και πολύ χρόνο. Στην ε, ε, παράγραφο 21 λοιπόν ε, δεν ενδείκνυται να συμπεριλάβουμε κάτι τέτοιο σχετικά με το σύστημα αδειοδότησης FLECT, ούτε ενδείκνυται όπως αναφέρεται στην παράγραφο 19 η Κομισιόν να παρεμβαίνει άμεσα στις υποθέσεις κυρίαρχου κράτους. Με τις διευκρινήσεις αυτές ε, κλείνοντας, ε, θέλω να ε, επικροτήσω την συμφωνία FLECT αυτήν, καθώς και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρία Πρόεδρο, προσβλέπω στην συζήτηση ε, για την σημαδιακή αυτή συμφωνία και να σας ευχαριστήσω για την σκληρή δουλειά και τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίσατε το σημαντικό αυτό θέμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την Επιτροπή Ανάπτυξης, ο κύριος Αρσένης για δύο λεπτά. Στο κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερως που συζητούμε εδώ το FLEGT, τη συμφωνία αυτή για την επιβολή δασική νομοθεσία διακυβέρνηση και το εμπόριο και αυτή την εθελοντική συμφωνία με την Ιδονησία, μια πολύ σημαντική χώρα που ε, έχει, κατέχει και ένα από τα σημαντικότερα τροπικά δάση στον κόσμο. Ένα τροπικό δάση που δυστυχώ όμω αποψηλώνεται με ραγδαία ταχύτητα. Η συμφωνία FLEGT είναι πολύ σημαντική γιατί μας δίνει ελπίδα ότι θα επιβραδυθεί κάπως ο ρυθμός αποψήλωσης αυτού του σημαντικού φυσικού πλούτου της Ινδονησίας. ο κύριος Ζαντό δέχτηκε τις τροπολογίες μου και θα ζητούσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη το Ινδονησιακό σύστημα διασφάλισης νομιμότητας της ξυλίας. Αν λειτουργεί σωστά, και τι προκλήσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε προκειμένου να λειτουργήσει σωστά για να τηρηθεί σωστά και η συμφωνία FLEGT. Θα ήθελα τώρα να επενέσω αυτή την συμφωνία FLECT, αυτό το πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό μηχανισμό. Γιατί σε αντίθεση με άλλες εμπορικές συμφωνίες ε, που έχουμε, η συμφωνία FLECT είναι μια διμερής εμπορική συμφωνία, πολύ σημαντική, που σέβεται όμως τα κυρίαρχα δικαιώματα των συμβαλωμένων μερών και εξασφαλίζει μεγάλη συμμετοχή των εμπλεκομένων. Και μάλιστα είναι παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες εμπορικές συμφωνίες που θα συνέψουμε με άλλους εταίρους μας. Θα ήθελα πάντως να πω και κάτι αρνητικό. Ως της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των δασών και την πράσινη βιβλό θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυστυχώς ε, παραμέλησε και αγνόησε όλες τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς την Πράσινη Βίβλο για την προστασία των δασών. Δυστυχώς ε, αδιαφόρησε πλήρως ε, όλες τις συστάσεις και τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί αυτή η περιφρόνηση. Σα ευχαριστώ. Τώρα έχουμε τους αγορητές των πολιτικών ομάδων για το ΕΛΚ. Τρία λεπτά. Έχετε το λόγο, συνάδελφε Κόστιγκερ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συζητάμε σήμερα μια σημαντική συμφωνία που αποτελεί σημαντικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής ε, για Βιωσιμότητα. Η Εθελοντική Συμφωνία εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με τρίτες χώρες έχει ε, πολλαπλή σημασία. Καταρχάς θέλουμε νόμιμη εκμετάλλευση των δασών σε κάθε κράτος μέλος με το οποίο συνάπτεται μια τέτοια συμφωνία. Επίσης θέλουμε βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων να ε, σεβόμαστε το περιβάλλον. Και τρίτον, με την Συμφωνία FLECT έχουμε πιο αποτελεσματική ανταγωνιστικότητα όσον αφορά τις εισαγωγές εξηλίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, η συμφωνία FLECT δεν είναι μια μεμονωμένη συμφωνία, είναι μέρος του αγώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, αποτρέψει την ε, παράνομη εκχέρσωση δασών και αποψήλωση δασών. με μεγάλη ταχύτητα γίνεται η αποψήλωση των δασών και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υπολογίζουν ότι κάθε χρόνο εισάγεται ξυλία, ε, παράνομη ξυλία αξίας 1,2 ε, δισεκατομμύριων ευρώ για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι πόροι αυτοί. Η συμφωνία λοιπόν ε, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ινδονησία αντιμετωπίζει ακριβώς το θέμα αυτό. Η η Ινδονησία προσλέπει σε ε, σύστημα πιστοποίησης. Εάν σκεφτούμε το δύσκολο σημείο κίνησης της ε, Ινδονησίας, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις πρόοδους που ήδη έχουν ε, σημειωθεί αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε διπλά μέτρα και σταθμά. Πολλά έχουν βελτιωθεί, ε, απομένουν όμως πολλά να γίνουν. Οι εργασίες τη συντονισία πάνω στη βιωσιμότητα στον δασικό τη τομέα θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα και να ε, επικροτηθούν. Γίνονται προσπάθειες ε, διαρθρωτικές και Πιστεύω ότι το ψήφισμα αναφέρει καλά τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε λάβει υπόψη μας στο κείμενο του κύκλους ενδιαφερομένων και επίσης έχουμε ασχοληθεί με τις συνέπειες στο περιβάλλον και τους ηθαγενείς χωρίς να ξεχάσουμε ότι η εθελοντική συμφωνία Εταιρική σχέση με την Ινδονησία ε, χρειάζεται τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να, ευχαριστώ όλους τους, να ευχαριστήσω όλους του συμμετέχοντες για την καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές. Ο κύριος Μάρτιν έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες και να ευχαριστήσω τον Γιάννη Ξαντό για το εξαιρετικό του έργο, όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά και για άλλε παρόμοιες συμφωνίε που είχαμε τη Λιβερία, Αφρικανική Δημοκρατία και το Καμέρον. Η αντιμετώπιση της παράνομη υλοτομίας ε, παγκοσμίω είναι μια τεράστια πρόκληση που θα πρέπει όμω να αναλάβουμε αν θέλουμε πραγματικά να σταματήσουμε την αποψήλωση, να προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα και να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Έχουμε ζωτικό ρόλο να διαδραματίσουμε σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Θα πρέπει το εμπόριό μας να στηρίζεται σε ηθικούς κανόνες. Δεν ε, θα πρέπει απλώ να λέμε δεν ξέρουμε την προέλευση της ξυλίας ε, και τι έγινε. Δεν πρέπει να επαναβαθούμε σε κάτι τέτοιο. Γιατί η δανεισή είναι σημαντικό ε, εξαγωγέα ξυλία προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει λοιπόν αυτό να γίνεται ει βάρο των δικαιωμάτων των γηγενών πληθυσμών που διαβιούν στο τροπικό δάσο ή ει βάρο τη ε, εις βάρος των δασών και εξαιτία αποψήλωση. Σίγουρα η Ιδονησία έχει από τα σημαντικότερα τροπικά δάση και αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις κυρίως εξαιτία της διαφθοράς. Η ιδονησιακή κυβέρνηση βέβαια και το αναγνωρίζουμε έκανε σοβαρή προσπάθεια για να καταπολεμήσει αυτή την παράνομη υλοτομία. Και χαίρομαι που θα γίνουν προσπάθειες για να ελεγχθούν οι εισαγωγές ξυλίας από την, από την Ινδονησία ώστε να αποφευθεί η εξαγωγή παράνομης ξυλίας και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, καλό θα ήταν να έχουμε έναν ενιαίο ε, online κανόνα παρακολούθησης, με χάρτη παρακολούθησης ε, της ξυλίας και καλό θα είναι τη χαρτογράφηση να μπορούν να την παρακολουθούν και, και οργανώσεις Τη κοινωνία των πολιτών. Επίση, οι άδειε που θα χορηγούνται θα πρέπει να είναι προσιτέ σε όλου. Και χαίρομαι για τα βήματα που έκανε η δανεισιακή κυβέρνηση που δείχνει συνεργάσιμο πνεύμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να ενθαρρύνω πάντως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ινδονησιακή Κυβέρνηση να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους για να στεφθεί με επιτυχία η συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπέρντερ έχει το λόγο για δύο λεπτά για την Άλντε. Για μας που προβληματόμαστε για την καταστροφή των τροπικών δασών, θα πρέπει να συγχαρούμε την ελληνική κυβέρνηση της προσπάθειας που καταβάλει να προχωρήσει με την προστασία των, της του ξυλοκομικού τομέα, τομέα της ξυλίας. Αυτή η θελοντική συμφωνία θα είναι σαφής ένδειξη ότι είμαστε αφοσιωμένοι στο να βοηθήσουμε και να ενθαρρύνουμε τέτοιες δράσεις είναι μια δέσμευση που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ελέγχει το πώς κόβεται η ξυλία από τα τροπικά δάση, να γίνεται με βιώσιμο τρόπο και ανιχνευσιμότητα. Μέχρι τώρα όλα πάνε καλά, μέχρι εδώ. Αλλά έχουμε τεράστιες ανησυχίες όσον αφορά το πώς ελέγχει τους δασικούς της πόρους η Ινδονησία στην περίπτωση του συστήματος αδειοδότησης που έχει. Ακολουθεί το σωστό δρόμο και αυτό είναι καλή πρόεδρος. Αλλά το SVLK ε, πρέπει να τα αντίμετρα κατά των παραβατών, να επιβάλλονται σοβαρές ποινές φυλάκισης και οικονομικές στους παραβάτες, πριν να μπορούμε να εμπιστευτούμε την εφαρμογή των μέτρων. Πρέπει να ξέρουμε ότι μόνο 10% των τροπικών κορμών της ε, Ινδονησίας έρχεται στην Ευρώπη. 90% εξάγεται προς χώρες με πολύ χαμηλές προδιαγραφές για το περιβάλλον, που έχουν διαφθορά. Και υπάρχει ατιμορρησία για το παράνομο εμπόριο όσον αφορά την, τα προϊόντα από τροπική ξυλία οι χώρε που έχουν τη φιλοσοφία του κέρδου σήμερα ε, ακολουθούν αυτό χωρί να νοιάζονται για το μέλλον. Λοιπόν, είναι θέμα για όλου μας η καταστροφή των δασών και κομπές αρνητικού και η απέτηση του, της δύση για την ξυλία και για το φινικέλαιο οδηγεί στην καταστροφή. Συμφωνώντας για αυτή τη συμφωνία είναι ένα μικρό βήμα προόδου προς ανιχνευσιμότητα, προς προστασία. Θα βοηθήσουμε τους Ινδονησίους να απαιτούν τα ίδια πρότυπα και από τους άλλους πελάτες. Αλλά μην πιστεύουμε ότι τελείωσε εδώ η δουλειά και ότι λυθήκαν τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για την ΚΟΕ το λόγο έχει ο κ. Μέρφυ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Ρόμπερτ Γκριν είπε ότι στη φύση δεν υπάρχουν ούτε αμοιβέ ούτε τιμωρίε, υπάρχουν συνέπειε. Και οι συνέπειε ε, τη αποψήλωση των δασών ε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνες για την βιοπικιλότητα, για τους ε, ηθαγενείς και για οποιονδήποτε μένει εδώ στον πλανήτη μας ε, και συχνά συνδέεται ε, με παρανομία και νομιμοποίηση παράνομων εισόδων. Η κλίμακα της αποψήλωσης των δασών στην Ινδονησία είναι τρομακριτή. Και η πολυεθνικές ε, σαν την Ferrero, την Unilever, την Estlé, ε, την Kraft, ε, την Hershey και την Wilmar International που κερδίζουν και που είναι υπεύθυνοι για αυτό. Και αν κάτι έχει αλλάξει αυτό οφείλεται στην πίεση του κοινού. Θέλω να σταματήσουμε την εισαγωγή παράνομης ξυλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι όμως υπέρ του εντοπισμού προβλημάτων στο πρόγραμμα και να μην θεωρήσει ότι το παρόν φλέκτε είναι η λύση για όλα ε, είναι απαραίτητο λοιπόν να γίνεται παρακολούθηση ε, και θα πρέπει οι ε, εταιρείε που συμμετέχουν στην ομοποίηση παράνομων εξόδων να ανακληθεί η άδειά τους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα έχουμε τη διαδικασία προσέλκυσης προσοχής του Προέδρου. Ο κ. Μπιέλαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την υπογραφή της ε, συμφωνίας αυτής με την Ινδονησία. Από άποψη ε, εμπορίας αποτελεί έκφραση της προσπάθειας να βελτιώσουμε, μια, ε, να βελτιώσουμε την κατάσταση και να ευνοήσουμε μια ισορροπημένη δασοκομεία σε, παγκόσμιο, σε παγκόσμια κλίμακα. Η Ινδονησία είναι πολύ σημαντικός εξαγωγέας ξυλίας, ενώ η ανεξέλεκτη η υλοτόμηση οδηγεί σε εξαφάνιση τροπικών δασών. Ελπίζω να, με τη συμφωνία αυτή να περιοριστούν οι πανταχού παρούσες διαφθορά και κερδοσκοπία στην Ινδονησία. Σας ευχαριστώ. Εκ νέου δίνω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Ποτότσνικ. Έχετε το λόγο. Thank you again. Ευχαριστώ και πάλι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους ευρωβουλευτές για την υποστήριξή τους και την έκφραση των ενισχυών τους σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας και την επιτόπια κατάσταση στην Ινδονησία. Ναι, ναι. Θα ήθελα να πω ότι σίγουρα η Ινδονησία είναι για μας πάρα πολύ σημαντική χώρα, γι' αυτό αξίζει κάθε προσπάθειας και με ιδιαίτερη χαρά συνάψαμε αυτή τη συμφωνία μετά από πολλές προσπάθειες που κάναμε. Γνωρίζουμε ότι η Δονησία εξακολουθεί να έχει κάποια προβλήματα και επίσης γνωρίζουμε ότι η χώρα αυτή προσπαθεί πάση θυσία, πασχίζει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Επίσης γνωρίζω ότι η εφαρμογή της συμφωνίας είναι πολύ σημαντική. Ε, με την εφαρμογή αυτή η Ινδονησία θα εφαρμόσει το ίδιο σύστημα εξαγωγών και σε άλλες ε, αγορές όπως αυτή της Κίνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά θα σας ενημερώσει με ιδιαίτερη χαρά για την πρόοδο εφαρμογής της συμφωνίας FLECT με την Ινδονησία και επίσης θα σας ενημερώνουμε για το κατά πόσο ε, λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα σημεία που αναφέρατε στο ψήφισμά σας επειδή μου θέσατε συγκεκριμένη ερώτηση για την ε, στρατηγική μας για τα δάση, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να ελέγξω τα στοιχεία που αναφέρετε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω πρόχειρα τα στοιχεία αυτά. Είμαι απροετοίμαστος και δεν θα ήθελα να δώσω ελαφρά την καρδία απαντήσει για τη στρατηγική μας για τα δάση. Θα ενημερωθώ και θα σα στείλω ακριβή απάντηση. Πάντως, όταν συζητούμε τα δάση, ε, συστηματικά και συνεχώς προσκρούμε στο επιχείρημα των κρατών μελών ότι αυτό το θέμα εμπίπτει στην επικουρικότητα και είμαστε υποχρεωμένοι να το λαμβάνουμε υπόψη. Πάντως σα διαβεβαιώ ότι θα το εξετάσω και θα σας στείλω απάντηση. Αν μου επιτρέπετε τώρα μια σύντομη ανακεφαλαίωση. Το μήνυμα που προέκυψε από τη συζήτηση ήταν σαφές και απερίφραστο. Αποκινούμε την Ινδονησία που είναι εταίρος μας και με τα κράτη-μέλη ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να φροντίσει ώστε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η συμφωνία. Έτσι θα φτάσουμε όλο και πιο κοντά στον απότερο σκοπό μας που είναι αναφυσβήτητα η βιώσιμη διαχείριση των ε, Ινδονησιακών δασών καθώς και η ευημερία των αυτόχθων πληθυσμών και όσων εξαρτώνται από τα τροπικά αυτά δάση. Σας ευχαριστώ. Λόγος στον εισηγητή για δύο λεπτά. Ο κύριος Σαντού έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ο στόχος αυτού του ψηφίσματος, όπως καταλάβατε πολύ καλά, δεν ήταν να προσθέσουμε νέους νομικούς όρους στη Συμφωνία Θελοντικής Εταιρικής Σχέσεως που ενεκρίθη. Υπάρχει μια συμφωνία, υπάρχουν νομικοί όροι που δεσμεύουν τα μέρη και στόχος του Κοινοβουλίου δεν ήταν να προσθέσει όρους και να δημιουργήσει νομική σύγχυση. Στόχος του Κοινοβουλίου ήταν προφανώς αυτός που ανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι. Δηλαδή να διαβεβαιωθούμε ότι οι άδειε φλεκτ που θα χορηγηθούν να εγγυώνται στους Ευρωπαίους πολίτες, στους καταναλωτές και στις Ευρωπαϊκές Αρχές ότι η ξυλία προέρχεται πράγματι από συστήματα βιώσιμα, ανοιχνεύσιμα και παρήχθησαν υπό καλές συνθήκες και επιστοποιήθηκαν και είναι νόμιμα διότι αν διαπιστώναμε κάποια δεδομένη στιγμή ότι οι άδειε φλεκτ που χορηγούνται δεν αντιστοιχούν σε, αυτό, σε αυτές τις προδιαγραφές, τότε όλος ο μηχανισμός φλεκτ θα υπονομευόταν εξού και η σημασία των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ευχαριστώντας σας για τη δέσμευση που αναλάβατε να έρθετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μας εξηγήσετε και να μας πείτε ποιες πρόοδοι επετέθησαν για, από πλευρά Ινδονησίας για το σύστημα επαλήθευση. Ε, ότι θέλετε να μας διαβεβαιώσετε πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως και εσείς από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από πλευρά των αρχών της Ινδονησίας όλοι μαζί συμβάλλουμε στην καλή ανάπτυξη της χώρας, την προστασία των δασών, την προστασία του κλίματος, την προστασία της βιοπικιλότητας και όλων των πληθυσμών που ζουν στα δάση ή που ζουν από τα δάση. Και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ έλαβα μια πρόταση ψηφίσματος, ολοκληρώθηκε η συζήτηση, η κοινή συζήτηση περατώθηκε, η ψηφοφορία επί του ψηφίσματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδονησίας θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Τελευταίο σημείο τη ημέρα διάταξη, η προφορική ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το αρχιπέλαγο των Σβάλμπαρντ και ε, τους αλληλευτικούς πόρους του αρχιπελάγους.